λόγο έχει ο εισηγητής ο κύριος Σοπφλίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τους σκιώδεις με τους οποίους συνεργάστηκα για αυτή την έκθεση, για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ήταν υποδειγματική η συνεργασία και μια ευχαριστή έκπληξη για μένα η ψηφοφορία στην ΑΦΚΟ πέτυχε ομοφωνία. Αυτή η ομοφωνία είναι σπάνια και αυτό από μόνο το αποτελεί ένα μήνυμα, μια ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεωρείται ε, εργαλείο κλειδί για το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα στην οποία βασίζεται είναι απλή οι πολίτες της Ευρώπης θα πρέπει να έχουν έναν τρόπο να ξεκινούν ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες για σημαντικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει η απομάκρυνση μεταξύ της Ευρώπης και των πολιτών της και το ECI είναι ένας τρόπος ε, να βελτιωθεί αυτό το πρόβλημα. Το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας των πολιτών δεν υπονομεύει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία που αποτελεί αξία θεμελιώδη οποιοδήποτε δημοκρατικού συστήματος και εμάς η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών όμως ενισχύει αυτή τη δημοκρατία με μια δράση των πολιτών που λειτουργεί παράλληλα με τα όσα πράττουμε εμείς. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν είναι κάποια άμεση δημοκρατία βέβαια που θα μπορούσε να λειτουργήσει στην αρχαία Ελλάδα, στα, ε, στις τη της αρχαίας Ελλάδας, αλλά δεν έχει νόημα όταν έχουμε να κάνουμε με εκατομμύρια πολίτες. Αυτό μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, είναι να κινητοποιήσει αρκετούς πολίτες συλλογικά για ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό το στοιχείο της κινητοποίησης δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Η διαδικασία συλλογής εκατομμύριων ε, ενό εκατομμυρίου υπογραφών εντό ενό έτου χρειάζεται ενθουσιασμό και δέσμευση για να γίνει κάτι σε πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Από αυτή την άποψη η πρωτοβουλία αυτή είναι ένας τρόπος συμμετοχής των πολιτών με τρόπο άμεσο, χωρίς δημεσολαβητή. Φυσικά πάντα θα υπάρχει κάποια ένταση μεταξύ της ε, αντιπροσωπευτικής πολιτικής ε, και των πολιτών. Η ιδέα ότι πολλοί πολίτες θα μπορούσαν να δράσουν μαζί για ένα ενίο ζήτημα προσθέτει κάτι καινούριο στην πολιτική παλέτα της Ευρώπης. Παρότι βέβαια πρέπει να σημειώνουμε ότι υπάρχει ίδια ω πολιτική δράση σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ε, εδώ η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών διαφοροποιείται από αυτήν ορισμένων κρατών μελών στο ότι η νομοθεσία ε, στα κράτη-μέλη ε, αρχικά ξεκινούσε από την Κομισιόν. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα και αλλάζει η ισορροπία διότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκινήσουν κάποια νομοθεσία. Αυτά θεωρητικά. Μέχρι σήμερα όμως ωστόσο δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι του μέσου αυτού. Πάνω από 50 πρωτοβουλίες οργανώθηκαν και καμία από αυτές δεν οδήγησε σε νομοθέτηση. Στις δικές μου διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών διέκρινα απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν χειρίστηκε τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που έλαβε. Υπήρξαν ε, διαμαρτυρίες για γραφειοκρατική καθυστέρηση και γενικά ενώ η Κομισιόν χρησιμοποίησε από νομική άψη πολύ σωστά το μέσο αυτό, έχει χάσει τον πολιτικό στόχο της εμπλοκής των πολιτών. Συνεπώς η έκθεσή μου εστιάζεται στην αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων και στην παρότρινση της Κομισιόν να ανταποκριθεί στη φωνή των πολιτών με μεγαλύτερη ευελιξία και ελπίζω ότι η υποσχεθήσα μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών θα τη μετατρέψει σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Φρανς Τίμερμαντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω τη σημερινή συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και χαιρετίζω την εξετρέψη Σόπφλιν. Επί αυτή τη βάση μπορούμε να συζητήσουμε κάτι το οποίο ε, είχε συζητηθεί και κατά την ακρόασή μου, άρα είναι κάτι που θα ήθελα ευχαριστώ να συζητήσουμε. Ω Επιτροπή, η Επιτροπή Juncker είπε ότι θα δράσει στα σημαντικά θέματα. Θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στα σημαντικά ζητήματα. Παράλληλα πρέπει να δούμε και πώς θα το κάνουμε. Και σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μπορεί να δώσει μια σημαντική συνεισφορά. Είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν οι πολίτες άμεσα να επηρεάσουν την πολιτική. Επιτρέπει στους πολίτες να να επηρεάσουν το ευρωπαϊκό θεματολόγιο και να προωθήσουν τα ζητήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Αποτελεί ένα έναυσμα πολιτικού διαλόγου. Όταν ήμουν στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, είχα συμμετάσχει και εγώ ίδιος σε πρωτοβουλίες πολιτών. Σήμερα, ως τμήμα των δραστηριοτήτων μου, ως αρμοδιότητά μου, είναι το να εξασφαλίζω ότι θα λειτουργούν καλύτερα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποια εμπειρία στον τομέα. Η Επιτροπή υπέβαλε μια έκθεση για τα πρώτα τρία χρόνια του θεσμού. Άρχισε να δείχνει κάποια αποτελέσματα. Καταγράφησαν 33 πρωτοβουλίε ε, για τι οποίε ε, συνελέγησαν υπογραφέ. Τρει ε, πρωτοβουλίε συγκέντρωσαν πάνω από ένα εκατομμύριο ε, ε, συμμετοχών και συνολικά πάνω από 6 εκατομμύρια πολιτών ε, υπέβαλαν δήλωση συμμετοχής. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο συμμετέσχουν σε μια προσπάθεια για κοινά ευρωπαϊκά ιδεώδια. Αυτό είναι μια πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία και για τη συμμετοχή του λαού υπό την έννοια της συμμετοχή του Δήμου στην αρχαία Ελλάδα στην έκθεση σας κύριε Σόφλιν υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία συμφωνούν με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα αναφέρω κάποια από τα μέτρα τα οποία ήδη ε, εφαρμόζονται. Η Επιτροπή ήδη έχει ένα σημείο επαφής στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν όλα τα, απευθυνθούν όλα τα ερωτήματα σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες. Επίσης δίνουμε άμεση βοήθεια στους ε, οργανωτές μόλις καταγραφεί μια πρωτοβουλία και δίνουμε πληροφορίες για νομικά θέματα και για τεχνικές ε, προϋποθέσεις. Πέραν των κανονισμών και διατάξεων επιτρέπουμε δωρεάν φιλοξενία στους διαμετακομιστές της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να επιτρέψουμε τη διευκόλυνση των απαιτήσεων για να μπορούν όλοι οι πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμά τους να υποβάλουν δήλωση συμμετοχή σε μια πρωτοβουλία πολιτών αν, αυτό, αν το επιθυμούν. Σήμερα θέλω να ακούσω με μεγάλη προσοχή τη δική σας αξιολόγηση για το πώς έχει λειτουργήσει αυτό το εργαλείο μέχρι τώρα και για το τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Η Επιτροπή σημειώνει το ότι προτείνεται μια αναθεώρηση της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και θα εξετάσουμε το πεδίο εφαρμογής μιας τέτοια αναθεώρησης. Θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία έχουν να πούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει ενεργά και σας ευχαριστούμε για αυτή τη συμμετοχή. Και προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Σέφλιν γιατί έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο με την ανάλυση που έκανε σχετικά με το πώς έχει υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μέχρι σήμερα σε όλες τις πολιτικές ομάδες και επιτροπές. Δεν προσπαθεί να κάνει μια πολιτικοποιημένη συζήτηση, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν κάποια σχέση με την Ευρώπη και με τον Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Διάλογο και πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει πιο εύκολη αυτή η προσπάθεια των πολιτών και πιο προσβάσιμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε. Η κυρία Κάφμαν από την Επιτροπή Δικαιοσύνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν. Θέλουμε και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα οικοδόμησης τη Ευρώπη. Αυτό είναι ακόμα και πιο σημαντικό όταν σκεφτόμαστε την πρωτοβουλία πολιτών. Πρέπει να λύσουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτέ οι πρωτοβουλίε πρέπει να κάνουμε περαιτέρω αλλαγέ, όχι απλώ ε, καλοπιστικές αλλά μία εκβάθρον αναδόμηση αυτής της οδηγίας. Πρέπει να έχει την υποστήριξή μας η πρωτοβουλία των πλοητών και να υπάρχει και η δυνατότητα τα, οι, αυτοί που κάνουν την πρωτοβουλία μετά την καταγραφή της πρωτοβουλίας να αποφασίσουν πότε θα ξεκινήσουν την ε, ε, τους και δεν θα πρέπει οι υπογραφές να συνδέονται με την εξακρίβωση της ταυτότητας αυτών που υπογράφουν. Πρέπει να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους νέους οι οποίοι θα πρέπει ήδη από τα 16 τους να μπορούν να υποστηρίσουν τις πρωτοβουλίες πολιτών. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι θετική. Είναι ελπίδα μου ότι η Κομισιόν πράγματι θα δεχτεί τις προτάσεις μας και θα τις εφαρμόσει ταχαίως και πρέπει από την παιδική ηλικία να ξεκινήσει αυτό το εργαλείο για να διαμορφώσει σωστούς πολίτες. Από την Επιτροπή αναφορών η κυρία Μπετσέρα Παστασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Η, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα εργαλείο συμμετοχής δημοκρατίας σε υπερεθνικό επίπεδο και έχει δημιουργηθεί για να επιτρέψει στους πολίτες να μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο με τι προτάσει του διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από τρία χρόνια που έχει εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, βλέπουμε ότι στην πράξη δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το ρυθμίσουμε με καλύτερο τρόπο και ζητάμε την Κομισιόν να τροποποιήσει την νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Πρέπει τα εργαλεία αυτά να εξυπηρετήσουν του στόχου που θέλουμε. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτών που κάνουν την πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Θα πρέπει να αναρμονιστούν οι εθνικέ προδιαγραφέ και να απλοποιηθεί η τεκμηρίωση, να υπάρξει ένα κοινό σύστημα για την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετέχουν, να έχουμε ευκαμψία για να υπάρχει ένα ευρύ διάστημα για τη συλλογή υπογραφών και να βελτιωθούν τα συστήματα πληροφορία Ανατολικής. Κυρίως όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να βοηθήσει να τροποποιηθεί το πρωτογενές δίκαιο. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ταχεία μεταρρύθμιση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, για να βελτιωθεί η πρωτοβουλία πολιτών, γιατί με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Περνάμε στις πολιτικές ομάδες από το ΕΛΚ, ο Τσάκη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό ασχοληθήκαν με το ζήτημα τρεις επιτροπές εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς ε, βλέπουμε τα πράγματα πιο θετικά όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά μέχρι στιγμής ε, τα τρία πρώτα χρόνια δεν έδειξαν ιδιαίτερα θετικά σημάδια και Χαιρόμαστε βέβαια που βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια συνένεση και ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών ε, συμμερίζομαι την άποψη αυτή. Οι πολίτες ε, είναι σημαντικό να νιώθουν ότι μπορούν να στραφούν στα θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλέ υποθέσει εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μάλιστα και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιοποιήσει αυτού τους κανόνε για το παραδεκτό ορισμένων πρωτοβολιών με κάποια μεγαλύτερη ευελιξία. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κύριε Τίμερμαν, θα μπορούσατε να δείξετε περισσότερη ευελιξία. Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη επιτυχία για τι ευρωπαϊκέ πρωτοβουλίε πολιτών στο μέλλον. Για την ομάδα των σοσιαλιστών η κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω αρχικά και εγώ τον εισηγητή, τον κύριο Σέπφλεν. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, γι' αυτό και ψηφίστηκε ομόφωνα. Η σκιωδής μας εισηγήτρια, η κυρία Κάφμαν, επίσης αξίζει τις ευχαριστίες μου για τις τεράστιες προσπάθειες που έχει καταβάλει για αυτό το θέμα εδώ και καιρό. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Τίμπερμαντς, εμείς σημειώσαμε με μεγάλη ευχαρίστηση τη δέσμευση που εκφράσατε εσείς εκ μέρους της Κομισιόν. Ωστόσο, αναμφίβολα, αυτά τα τρία πρώτα έτη εμφανίστηκαν πολλές δυσκολίες για την πρακτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής. Πιο συγκεκριμένα θέλω να υπενθυμίσω ότι πρέπει να γίνει πιο σαφής η διαδικασία, όχι η διαδικασία εγγραφής, και καταχώρησης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούν συγκεκριμένα ομάδες πολιτών κατά πόσο υπάρχει τέτοια δυνατότητα ε, για να προσφέρουν κάποια πρωτοβουλία που να συνάδει με τις συνθήκες. Μετά πρέπει να διευκολύνουμε τη συγκέντρωση των υπογραφών και εμεί έχουμε προτείνει μια σειρά ε, ώστε να διευκολυνθούν και να απλουστευτούν ε, η συλλογή των υπογραφών και να ευνοηθεί η συμμετοχή των πολιτών, οι χρόνη, οι συνθήκες ε, υποβολής, ε, η χρόνη από το τέλος της εγγραφής και την έναρξη της συλλογής, οι online υπογραφές, πολλά στοιχεία. Αλλά μετά υπάρχει και κάτι πολύ βασικό. Η πρόταση της Κομισιόν και από αυτού εμείς ε, θέλουμε μεγαλύτερη δέσμευση τη Κομισιόν. Αν υπάρχει εγγραφή και υπάρχουν και υπογραφές, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια πρόταση, να ακολουθήσει κάποια πρόταση εκ μέρου των θεσμών. Ευχαριστώ. Εκ μέρου του ECR, ο κύριος Ουζαντζόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σέφλιν όχι μόνο γιατί κατόρθωσε να δημιουργήσει συνένεση, αλλά κυρίως διότι εξ αρχής υπέβαλε αυτή την έκθεση με στόχο την αναζωογόνηση αυτού του θεσμού. Οι προτάσεις του αποσκοπούν στο να εξελιχθούν οι γραφειοκρατικοί φραγμοί και να εξασφαλιστούν όλα όσα θα συνεισφέρουν ε, στην καλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Υπάρχουν κάποια λεπτά θέματα στην έκθεση που πρέπει να συζητήσουμε. Ε, καταρχήν, ρωτά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς και πότε θα μπορέσει να μειώσει ε, κάποιες αυθαίρετες ενεργειές της. Η πρωτοβουλία «Ένας από εμά απερίφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά την ευρεία στήριξη που είχε και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Πιστεύω ότι μια πρωτοβουλία που έχει λάβει την υποστήριξη με τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών θα πρέπει να λάβει κάποια συνέχεια με νομοθετική πρωτοβουλία. Θα ήθελα λοιπόν να, να δω πώς θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την έκκληση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια νέα τροποποίηση του κανονισμού. Και ευχαριστώ τον κύριο Σιγητή για την εξαιρετική έκθεση που έχει υποβάλει. Από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Θέλουμε να είναι ένα πραγματικό δικαίωμα, όχι μόνο στα χαρτιά ένα δικαίωμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρους ομάδας των Φιλελευθέρων, ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα καινοτόμο μέσο της συνθήκης Λισαβόνας ε, για να ε, ε, βελτιστοποιήσει τη ε, δημοκρατία στην Ευρώπη. Ποιο δεν θέλει να συμμετέχουν οι πολίτες φυσικά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ε, αξιολογούμε ε, μετά από τόσα χρόνια τη λειτουργία χωρίς να αμφισβητούμε την αρχή. Πολλές πρωτοβουλίες έχουν προσκρούσει σε διάφορα εμπόδια με αποτέλεσμα τελικά να εγκαταλειφθούν τα έργα. Θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον εισηγητή και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων η οποία ομόφωνα βοήθησε στη βελτίωση ε, της πρωτοβουλίας. Εμείς υποστηρίζουμε τις προτάσεις ελάμφρυσης της διαδικασίας και παράλληλα μας φαίνεται σοφό η Επιτροπή αυτή να ασχοληθεί με τα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμόδιότητές της και να αναθέσει τα υπόλοιπα στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Εάν συμμεριστούμε τις απόψεις του εισηγητή, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε να διευκρινίζουμε ως ομάδα ALDE ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δέχεται και πρωτοβουλίες που αφορούν πρωτεύουν δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή την άποψη παραβλέπουμε ότι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά περιορίζεται από τις συνθήκες. Η Επιτροπή, έχοντας ε, το δικαίωμα πρωτοβουλίας για αλλαγή της συνθήκες, ε, είναι έτσι θεματοφύλακας και των προτάσεων των πολιτών. Για αυτό το σκοπό, εμείς μαζί με την ομάδα των Πρασίνων υποβάλαμε μια τροπολογία με την οποία ε, θα θέλαμε η πρωτοβουλία των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών να μπορεί να ασχοληθεί και με ζητήματα ε, των συνθήκων για την ομάδα ε, Γκουε η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ. Η Ένωση ανακάλυψε τη συμμετοχική δημοκρατία μετά από μια κρίση. Η Βόρεια Ιρλανδία με τη συνθήκη της Νίκαιας και τώρα με την πρωτοβουλία των πολιτών δίνουμε μια απάντηση σε αυτή την κρίση. Σήμερα η κρίση έχει επιδεινωθεί και η συμμετοχική δημοκρατία ε, πεθαίνει καμία πρωτοβουλία με απερκή αριθμό ε, υπογραφών δεν ακολουθήθηκε από κάποια νομική δράση. Δεν είναι τέλεια η έκθεση Σέπφλιν, δεν επιτρέπει αλλαγή των συνθήκων, αλλά ψηφίστηκε ομόφωνα από την Επιτροπή ΑΦΚΟ, διότι διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την νομική παρακολούθηση των πρωτοβουλειών. Εγώ θα ήθελα επίσημα να ζητήσω από αυτό το Κοινοβούλιο να καταψηφίσει την τροπολογία 4 της παραγράφου 3 με την οποία ε, θα ευνοχιστεί ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Το ζητώ από σοσιαλιστές που την επέβαλαν. Η τροπολογία αυτή ζητά από την Κομισιόν να προτείνει νομοθετική ε, πράξη μόνο αφού έχει δοθεί θετική γνωμοδότηση. Μέχρι σήμερα 29 πρωτοβουλίες από τις 49 έγιναν δεκτές, οι τρεις ε, ε, ε, επέτυχαν τις υπογραφές και μόνο το δικαίωμα στο νερό έλαβε κάποια θετική γνωμοδότηση. Καμία δεν μεταφράστηκε σε νομοθεσία. Η Επίτροπος Μάλμστρεμ απάντησε στις αναφορές κατά του TTIP δεν λαμβάνω εντολή από, τον Ευρωπαϊκό, από τους λαούς της Ευρώπης. Θα ήθελα να μας πει και αυτή η κυρία Αντιπρόεδρε Τίμερμανς και από και εσείς κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς από ποιον έχει λάβει σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν εντολή. Ευχαριστώ. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει ο κύριος Τερικάβρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα των Πρασίνων Ελεύθερη Συμμαχία έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με μεγάλο ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση πρωτοβουλία πολιτών, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό διορθωτικό εργαλείο ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να φέρει πιο κοντά τους πολίτες στα θεσμικά όργανα. Και έτσι μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η απόσταση και η αντίληψη της ε, ε, υπεροψίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτή του φίλου μας, του κ. Σέφλιν, είναι πάρα πολύ θετική. Είναι γεγονός ότι ενεκρίθη ομόφωνα στην Επιτροπή μας. <clears throat> Παρά της θετικής αυτής άποψης πρέπει να αναφέρω κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει τύχει περισσότερης προσοχής και περισσότερου θάρρους από μας. Πρόκειται για την απαραίτητη τροποποίηση της παρακολούθησης οποιασδήποτε επιτυχούς πρωτοβουλίας πολιτών μετά από την υποβολή τους. Με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε και τις ευρωπαϊκές αυτές πρωτοβουλίες. Μια τέτοια συνέχεια σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα και να προετοιμάσουμε τις νομικές πράξεις, νομοθετικές πράξεις επί τη βάση των κανόνων της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν και οι οποίες κατά την άποψή μου δεν εκφράσουν σαφώς τον στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Για να είμαι τελείως ειλικρινής πρέπει να πω ότι αυτές οι τροπολογίες σε κάποιο βαθμό πηγαίνουν αντίρροπα από αυτό το οποίο πρέπει να επιτύχουν οι πρωτοβουλίε πολιτών. Γι' αυτό έχουμε παρουσιάσει και τι δικέ μα τροπολογίε ω ομάδα των Πρασίνων για να δώσουμε στην Κομισιόν και το Κοινοβούλιο την ευκαιρία να διαδραματίσουν ένα πιο μεγάλο και πιο σημαντικό ρόλο προ την κατεύθυνση τη υποστήριξη των δημοκρατικών οθήσεων από του πολίτες που θέλουν μια ισχυρότερη και πιο δίκαιη Ευρώπη. Ελπίζω ότι οι τροπολογίε μα μπορούν να αντλήσουν μια πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα, λέει ο Πρόεδρο. Το λόγο για την Ευρώπη των Εθνών και τη Δημοκρατία και των Ελευθεριών, ε, ο κ. Καστάλντο. Πολλέ προσδοκίε, ε, με λίγα λόγια, για αυτό το κύριο εργαλείο άμεση δημοκρατία σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ένα βασικό πυλώνα για το κίνημα των Πέντε Αστέρων. Οι συνάδελφοι υπενθύμησαν το πλήθο ε, το πρωτοβουλίο που ξεκίνησε και μόνο τρει έγιναν αποδεκτέ λόγω γραφειοκρατίας, έλλειψης ενημέρωσης, έλλειψης ε, ομοιομορφίας, ομοιόμορφης αντιμετώπισης μεταξύ κρατών μελών και για τη συλλογή υπογραφών και για την νομική βάση. Αυτή η έκθεση δίνει κάποιες απαντήσεις μεν ε, για πρακτικά θέματα και συγχαίρω τον ε, κύριο εισηγητή, τον κύριο Σέπφλιν. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε πιο σημαντικά βήματα, πολιτικά βήματα να επιλύσουμε τη σύγκρουση συμφερόντων με την Κομισιόν όπου από τη μια μεριά ελέγχει το, το παραδεκτό και από την άλλη αποφασίζει αν θα νομοθετήσει ή όχι βάση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας ε, αφού ολοκληρωθεί η διαδρομή της δεν μπορεί αυτό να γίνεται προαιρετικά. Πρέπει να είναι υποχρέωση για να είναι αξιόπιστοι οι θεσμοί και να πλησιάσουν τους πολίτες. Δεν μπορούμε να αναιρούμε τις προσπαθίες τους εδώ στην έδρα της Δημοκρατίας. Πρέπει να διασώσουμε αυτή τη βούληση και να ε, την ενισχύσουμε να επιτρέπει και αλλαγή των συνθήκων να σταματήσουμε αυτή την απραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δοθεί μια όθηση από τους πολίτες ώστε ε, να γίνει πραγματικότητα το όνειρο των προπατόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν των όσων επιθυμεί η κυρία Μάλμστρομ. Ευχαριστώ. Για την Ευρώπη των Εθνών και των Ελευθεριών, ο κύριος Άνεμανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αν είχε λειτουργήσει στην εντέλεια αυτό το μέτρο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών, πάλι θα διαπιστώναμε ένα δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρώπη. Κάποια από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία πλήττουν τους πολίτες ε, προβάλλονται μέσω των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλίων Πολιτών αλλά δυστυχώς οι μόνες πρωτοβουλίες που κατάφεραν να περάσουν από τη γραφειοκρατία είναι ελάχιστες. Και δεν ε, καταφέραμε να έχουμε νομοθετικές προτάσεις ως αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να συνεχίσει με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες στις ε, ε, πρωτοβουλίες αυτές. Ευχαριστούμε κύριε Άνεμανς, ο συνάδελφος Μπαλτσό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο που εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς είναι πολύ αδύναμο εργαλείο χρειάζονται ένα εκατομμύριο υπογραφές και το μόνο που μπορεί να επιτύχει κανείς είναι σύνταξη μιας πρότασης από την Επιτροπή. 51 πρωτοβουλίες ε, προέκυψαν, μόνο τρεις ήταν παραδεκτές και δεν ακολούθησε καμία νομοθετική πρωτοβουλία. Τώρα προσπαθεί ο εισηγητή να υποβάλει κάποιες τροπολογίε για βελτίωση του συστήματος, αλλά δεν βλέπουμε τρόπο βελτίωση. Αν δούμε την κρίση σχετικά με τους πρόσφυγες, βλέπουμε ότι η πολιτική ελίτ στην Ευρώπη είναι πολύ απομακρυσμένη από τους πολίτες, από το επίπεδο των απλών πολιτών. Υπάρχουν πάρα πολλέ και έρευνε που δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση Υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ πολιτών και πολιτικής ελίτ. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό δημοψήφισμα. Αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία. Αυτό θα έπρεπε να εισαγάγουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστούμε κύριε Μπαλτσό. Από τη συνάδελφο Κόμπερν δέχεστε μια ερώτηση κύριε Κόμπερν. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλτσό και κύριε Πρόεδρε. Μια απλή ερώτηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Συμφωνείτε μαζί μου ότι αν οι άνθρωποι σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο δεν μπορούν να υποχρεώσουν να προωθηθεί μια πρωτοβουλία από αυτό εδώ το κοινοβούλιο, πώς φαντάζεστε ότι θα μπορούσαν οι πολίτες να πράξουν το ίδιο. Όλο αυτό είναι χάσιμο χρόνο. Συμφωνείτε μαζί μου κύριε Κύριος Βάλτσο, Κοιτάξτε, αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, λέτε ότι ουσιαστικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε κάποια πράγματα μέσα το κοινοβούλιο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να δίνουμε την ίδια επιλογή στους πολίτες. Όχι, δεν είναι χάσιμο χρόνο αν χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο το οποίο θα παρέχει ένα σαφές πλαίσιο το οποίο θα λειτουργεί διαφορετικό από τη σημερινή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών γιατί νομίζω στη δική σας χώρα ε, υπάρχει ε, το δημοψήφισμα οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο παρόμοιο με αυτό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευχαριστούμε κύριε Μπαλτσού Η κυρία Σουίτσα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Με τη συνθήκη της Λισαβόνας υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και αντίθετα από τον συναδελφό εγώ θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που βοηθά τους πολίτες μας ε, να συμμετέχουν σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Ξέρω ότι μόνο τρεις ε, έφτασαν σε κάποιο πέρας, αλλά καμία δεν ακολουθήθηκε από κάποια νομοθετική πράξη. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Σόπφλιν ε, για τις προσπάθειες που κατέβαλε για αυτή την έκθεση. Πιστεύω και ελπίζω η Κομισιόν να γίνει πιο δραστήρια, να βοηθήσει στη συλλογή υπογραφών με ευκολότερο τρόπο, να βοηθήσει στην ταχύτερη εγγραφή τους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δοθούν κίνητρα στην Κομισιόν να δράσει. Πιστεύω ότι το εργαλείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά Πρέπει να ευθυγραμμίσουμε και τις εθνικές νομοθεσίες ε, με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ θετικό εργαλείο. Ευχαριστούμε κυρία Σνίτσα και κυρία Ταπαντέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η άμεση δημοκρατία, σύμφωνα με το μοντέλο της Αρχαίας Αθήνας, ε, δεν είναι ε, μόνο ένα αρχαίο σύστημα, είναι και ένα σύγχρονο σύστημα που μπορεί να επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Κατετέθησαν 51 πρωτοβουλίες και πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες αγωνίστηκαν για να αλλάξουν την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει όμως να έχουμε μια εσφαλμένη εικόνα. Μόνο τρεις πρωτοβουλίες θεωρήθηκαν παραδεκτές και καμία δεν οδήγησε σε νομοθετική πρωτοβουλία. Τώρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το ότι πρέπει να βελτιώσουμε την επιτυχία αυτού του μέτρου. Και τι μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα συλλογής υπογραφών online και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες σε υψηλότερο επίπεδο. Στους νέους θα βρούμε μια λύση γιατί οι νέοι έχουν επίγνωση της κοινωνίας στην οποία ζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι νομίζουμε και θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε μια ευχάριστη έκπληξη σε ένα δώρο το οποίο θα κάνουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό προτείνω να μειώσουμε την ηλικία των συμμετεχόντων από 18 σε 16 ετών για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχημένα μέτρα στο μέλλον χρησιμοποιώντας τους νέους και όλο το δυναμικό το οποίο μπορούν οι νέοι να δώσουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ταπρατέλ. Δεν βλέπω καμία γαλάζια κάρτα. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που θεσπίστηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί σημαντική κατάκτηση των λαών της Ευρώπης και ενισχύει τη συμμετοχική δημοκρατία στο πλαίσιο της Ένωσης ταυτόχρονα αποτελεί μια μορφή πλατιά συνεργασία των πολιτών και των κινημάτων σε πανενωσιακό επίπεδο ενισχύοντα έτσι του δεσμού αλληλεγγύη και κοινωνική δράση. Ω συντονιστή του ecr στην επιτροπή αναφορών έχω επανειλημμένα επισημάνει τι αδυναμίες του εφιστάμενου νομικού πλαισίου του κανονισμού 1179 του δύο που πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου πρώτον για να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών ιδίως στην παρούσα περίοδο της οικονομικής κρίσης; δεύτερον προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα. πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούν ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών συνιστά πρωτογενή άσκηση της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους πολίτες και τα κινήματα του ευρωπαϊκού νότου για τη δημιουργία ενός πλατιού μετώπου ενάντια στη λιτότητα και στη φτώχεια ενάντια στην ασυδοσία της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και της ευρώπης των τραπεζών και εμείς οι αντιμνημονιακοί πολίτες θα αναλάβουμε σχετική πρωτοβουλία στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Ο κύριος Ντιρόν για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Τίμερμαν, στο 2009 οι Συνδίκες της Λισαβόνας προσπάθησαν να δημιουργήσει άμεσο σύνδεσμο μεταξύ πολιτών και Ευρώπης. Η πραγματικότητα είναι ότι απέτυχε πλήρως. Αναφέρθηκε προηγουμένως υπήρξαν 51 ή μάλλον 53 πρωτοβουλίες πολιτών με, τα, με τις τελευταίες που κατετέθησαν. Τρεις είχαν πάνω από ένα εκατομμύριο πολιτών που τις υποστήριζαν και δεν προήλθε από όλα αυτά τίποτα. Εγώ έχω πρόβλημα. Γιατί οι πολίτες δεν είναι πιο χαζοί από τους ευρωβουλευτές ή τους επιτρόπους. Και κάνουν κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Χρειάζονται τεράστια κινητοποίηση, λεφτά, ενέργεια που επενδύουν οι πολίτες αυτές τις εκστατείες και βλέπουν ότι τίποτα δεν βγαίνει από όλα αυτά και από τις πολλές πρωτοβουλίες έχουμε κατέβει τώρα πια σε ένα ασήμαντο και γελίο αριθμό πρωτοβουλειών. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Υπάρχει μια εναλλακτική δυνατότητα. Ή θα κάνετε τις απαραίτητες νομοθετικές ε, πράξεις. Διακόπτει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό κύριο Σβέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σόπλεν για την τόσο καλή έκθεσή του για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Δίνει τη δυνατότητα στου πολίτε να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Φυσικά υπάρχουν προποθέσει. Η έκθεση αυτή προσπαθεί να βελτιώσει αυτό το τόσο πρωτότυπο και σημαντικό εργαλείο ευρωπαϊκή δημοκρατία. Να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα, να δημιουργηθούν οι κατάλληλε συνθήκες ώστε να μπορεί να ευδοκιμήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών έχει μετά από τρία χρόνια ε, γίνει αντικείμενο πάνω από 50 πρωτοβουλειών, αλλά μόνο τρεις έχουν ξεπεράσει το αναπαραίτητο αριθμό ε, υπογραφών και καμία τελικά δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί. Αυτό δεν είναι υπέρ της ε, δημοκρατίας, δείχνει τις ατέλειες της δημοκρατίας. Πιστεύω όμως ότι αυτές οι μορφές άμεσης δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάνουν πιο ζωτική την ευρωπαϊκή δημοκρατία και βοηθούν να υπάρξει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω την έκκληση που περιέχεται στην έκθεση Σέπλιν, οι φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τι πρωτοβουλίε πολιτών και έτσι να κερδίσουν την πρωτοβουλία, την, ε, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Γιατί χωρί του πολίτε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Τσβέρ. Για ένα λεπτό η κυρία Μίτσι. Sir President, the European Citizens Initiative, Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι το πρώτο τέτοιο εργαλείο το οποίο δίνει στους πολίτες δυνατότητα να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Πρέπει λοιπόν να τεθεί στο ίδιο επίπεδο αυτή η δυνατότητα πρωτοβουλίας με τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν που είναι θεσμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά φαίνεται πάρα πολύ απόμακρα. Με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια άμεση έκκληση που γίνεται από τους πολίτες και μπορεί να τους φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη. Αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από την πρωτοβουλία πολιτών. Ήταν φρούδα όμως όπως έδειξε η πραγματικότητα. Υπήρξαν, ε, υπήρξαν σκικαίωνας από γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια που δεν επέτρεψαν στους πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο και να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να τροποποιήσουμε τους κανόνες για την πρωτοβουλία πολιτών για να γίνει πιο φιλική προς τους πολίτες και να μπορεί να αναπτύξει όλες τις δυνατότητές της. Ευχαριστώ κύριε Μίτση. Ο κύριο Γκέρι και για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε όταν στην ε, Γερμανία ε, πηγαίνω από τη μία πόλη στην άλλη, ακούω πολλές φορές ε, ότι εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ενδιαφερόμαστε για τους απλούς πολίτες. Η Ευρώπη χρειάζεται την άμεση δημοκρατία. Η Ευρώπη χρειάζεται να κινητοποιήσει τους πολίτες άμεσα. Πρέπει να τολμήσουμε τη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που να μην είναι γραφειοκρατική και να είναι αποτελεσματική. Δεν μπορούν οι πολίτες να ασχολούνται με κάτι από το οποίο δεν προκύπτει τελικά τίποτα. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να τολμήσουμε τη δημοκρατία και να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό κίνημα που θα ενισχύει τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Γκίκολτ. Ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Τσαμπόρσκα. Ďakujem, pán predseda som Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που ο εισηγητής κύριε Σέπφλινγκ ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στην έκθεσή του. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ένα πραγματικά ευρωπαϊκό δημοκρατικό εργαλείο. Υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν εκρίθησαν παραδεκτές. Υπήρξαν και πρωτοβουλίες όπως η, ε, ένας από εμά, στις οποίες δεν δόθηκε συνέχεια. Δόθηκε η ευκαιρία στην Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις πρωτοβουλίες των πολιτών και θα πρέπει στο μέλλον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να βοηθήσουν τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρσκα. Έχω περισσότερους ομιλητές που ζητούν το λόγο. Θα περιοριστούμε λοιπόν σε ένα ομιλητή αναπολιτική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τρία συμπεράσματα μπορούμε να εξαγάγουμε από αυτή τη συζήτηση. Πρώτον, η πρωτοβουλία πολιτών είναι πολύ σημαντική για τη δημοκρατική συμμετοχή. Δεύτερον, η τωρινή νομοθεσία δεν λειτουργεί. Τρίτον, πρέπει να τη βελτιώσουμε. Μέχρι εδώ συμφωνούμε όλοι. Θα ήθελα να πω στον κύριο Τίμερμαν ότι για μένα υπάρχει μια λύση η οποία θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα από πολιτική έποψη για να κάνουμε τη μεταρρύθμιση μετά τη πρωτοβουλία πολιτών. Δηλαδή, για τι πρωτοβουλίε που φτάνουν το 1 εκατομμύριο υπογραφών αλλά που δεν θεωρούνται παραδεκτές για λόγους αρμοδιοτήτων ή για άλλους νομικούς λόγους να τους δίδεται μια θεσμική απάντηση, να καθορίζεται κάτι τέτοιο. Να μην αφήνουμε να περάσει τη μια πρωτοβουλία που έχει τόση μεγάλη ικανότητα συνάθρησης ανθρώπων για λόγους νομικούς ή τυπικούς και να μην μπορεί να ετύχει μια συνέχεια προτείνω λοιπόν η Κομισιόν να απαντά επισήμω, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραπέμψει σε άλλε νομικέ διαδικασίε ή σε άλλε πρωτοβουλίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χαουρεγγί. Ο κύριο Σκρικ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Τόσες φορές συζητάμε επίσημα και ανεπίσημα το ίδιο θέμα. Από το 2012 έχουμε αυτό το μέσο στην ευρωπαϊκή πολιτική και κάποιες ε, πρωτοβουλίες ε, επιτυχής ε, κατέδειξαν τις αποτυχίες μας γιατί δεν καταλήξαμε σε καμία νομοθεσία. Οπότε κάνω μια έκκληση εδώ να κολοσορίσουμε αυτή την πρόταση της, του εισηγητή για καλύτερη προσβασιμότητα του μέσου, αλλά αυτό δεν αρκεί. Κύριε Επίτροπε, εξηγήστε στους πολίτες την έλλειψη διαφάνειας επί του θέματος. Πώς γίνεται ο θεσμός που είναι αρμόδιος γι' αυτό να ελέγχει και το παραδεκτό και όχι να κάνει αυτό τον έλεγχο κάποιος ουδέτερος οργανισμούς. Έχει αιτιολογήσει επαρκώς τις απορρίψεις των ε, το στο παρελθόν ε, η Επιτροπή ε, που ξέρουμε ότι έχει του σωστού λόγου. Ή μήπω είναι ζήτημα πολιτική ορθότητα όλο αυτό, όταν έχουμε σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτε που λένε ε, να μην ε, σκοτώνουμε μωρά πριν από τη φυσική γέννα ή δεν μας αρέσει πια αυτό. Θα, ε, πώς θα γίνει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στο NSA. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φερέρα έχει το λόγο. Ο κύριος Φερέρα, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να αναφέρω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει την εντύπωση ότι είναι δημοκρατική, αλλά δεν είναι σύμμορφη με τη θέληση των λαών. Η λεγόμενη πρωτοβουλία πολιτών είναι μια πρωτοβουλία πεδαριώδης για να, να νομιμοποιηθεί ένα οικοδόμημα το οποίο είναι βαθιά αντιδημοκρατικό. Η συνθήκη της Λισαβόνας το έκανε αυτό για να δώσει την εντύπωση ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια συμμετοχή των λαών. Αλλά η συνθήκη αυτή έγινε δεκτή χωρίς δημοψηφίσματα, χωρίς την θέληση των πολιτών. Μετά από έξι χρόνια λοιπόν που έχουν περάσει, είναι φανερό ότι έχει αχυρώθηση τον εαυτό του αυτό το εργαλείο που υποτίθεται είναι τρόπο συμμετοχή. Μόνο τρει πρωτοβουλίε έφτασαν τα άκαμπτα όρια του ενό εκατομμυρίου για να θεωρηθούν ότι είναι συμμετοχή πολιτών και μετά η Κομισιόν τη ακύρωσε όπω αυτή για το νερό, το οποίο πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα. Ο κύριος Σόλτες έχει το λόγο. Σόλτες. Eh, eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα εργαλείο άσκησης άμεσης δημοκρατίας. Έχουν ε, ήδη ε, γίνει πολλές πρωτοβουλίες πολιτών χωρίς αποτέλεσμα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε καμία πρωτοβουλία και αυτό δημιούργησε σύγχυση και απογοήτευση μεταξύ των πολιτών. Θα πρέπει να ακολουθείται από κάτι συγκεκριμένο η πρωτοβουλία πολιτών. Αυτό υπάρχει στη νομοθεσία σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών και θα έπρεπε να εφαρμόζεται κιόλα. Ήδη συζητήσαμε το θέμα του παραδεκτού. Θα πρέπει και τα κριτήρια να προσαρμοστούν και οι κανόνες να είναι σαφείς και αποτελεσματικοί. Αν οι κανόνες δεν είναι σαφείς, δεν θα επιτύχει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, θα παραμείνει μια ψευδέστηση. Ευχαριστούμε κύριε Σόλτες, συνάδελφος Άρνολτ. The word citizens initiative η λέξη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών φαίνεται εξαιρετική ιδέα της περισσότερης δημοκρατίας, της μεγαλύτερης δύναμης που προκύπτει από τους ε, πολιτικούς, τους οποίους δεν εμπιστεύονται οι πολίτες, ε, ε, εξουσίες η οποία επιστρέφει στους πολίτες. Ακούγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά από όλες τις πρωτοβουλίες μόνο τρεις κρίθησαν παραδέκτες από τις 51 που υπευλήθησαν θα ήταν δημοκρατικό δικαίωμα των ε, πολιτών ε, να επιτυγχάνουν κάτι με τις υπογραφές τους. Σήμερα χρειάστηκε να ταξιδέψω μέσω της Ελβετίας και σκέφτηκα ότι η Ελβετία δίνει το καλό παράδειγμα γιατί οι πολίτες μπορούν με ένα δημοψήφισμα να συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Καταπληκτικό παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας. Η Ελβετία μας δίνει το καλό παράδειγμα και πιστεύω ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διδαχθούν από το παράδειγμα της Ελβετίας. Ευχαριστούμε κύριε Άρνετ και κλείνοντα τη διαδικασία διάρκεια ο συνάδελφο Σόμπερμαγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι καλή ιδέα η ιδέα της πρωτοβουλίας πολιτών, αλλά είναι πολλά που μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν λειτουργήσει. Έχουμε 53 πρωτοβουλίες από τις οποίες καμιά τελικά δεν έχει υλοποιηθεί και δεν έχει τύχει διαδικασίες επεξεργασίας. Ούτε αυτή για την TTIP. Πώς ε, πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το σύστημα και να υπάρχει μια φιλική προς τον πολίτη ε, διαδικασία για την πρωτοβουλία πολιτών. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να δώσουμε δημοκρατικό χώρο ε, συζήτησης και δράσης των πολιτών. Γιατί αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής με τη μορφή που έχει είναι απλώς ένα πλασέμπο. Είναι κάτι το οποίο δίνει την εντύπωση της δημοκρατίας χωρίς να την εξασφαλίζει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Όμπερ Μάιερ. Τώρα για την Κομισιόν έχει το λόγο ο κύριος Τίμερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο να ξαναπώ αυτό που είπα προηγουμένως. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνεργαστεί πολύ στενά με τον κύριο Σέφλιν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό μπορούμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις ε, βελτιώσεις που προτείνει η έκθεσή του για την πρωτοβουλία πολιτών. Προσβλέπω λοιπόν σε μια ενισχυμένη συνεργασία μαζί σας, ώστε να μπορέσουμε πράγματι να βελτιώσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Για να το κάνουμε αυτό λοιπόν θα πρέπει να επανέλθουμε στον κανονισμό, αλλά η Κομισιόν δεν θα παραμείνει άτολμη ενώπιον αυτής της ανάγκης να υπάρξουν τροποποιήσεις. Συγχρόνως όμως μπορώ να σας πω ότι μπορεί να μετατρέψετε την πρωτοβουλία σε κάτι το οποίο δεν θα σας αρέσει και μετά να το επικρίνετε. Αλλά βασίζεται πάνω στη συνθήκη αυτή η πρωτοβουλία πολιτών. Είναι κάτι το οποίο το ενέκριναν όλα τα κράτη-μέλη και το κύριο αναστατικά κοινό Μπορεί να ήταν ωραίο να ξεπεράσουμε αυτά που λένε οι συνθήκες, αλλά εμεί δεν μπορούμε, γιατί η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακα των συνθήκων και οι κανόνε λένε ότι η πρωτοβουλία πολιτών είναι ένα εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών σε διάλογο. Δεν είναι μια πρωτοβουλία που δίνει νομοθετική πρωτοβουλία στους πολίτες. Αν δεν σας ικανοποιεί λοιπόν αυτή η ρύθμιση, εντάξει, αλλά δεν φταίει αυτή η ρύθμιση ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ο στόχος της είναι να είναι μια προσθήκη στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία για να εξασφαλίσει ότι θα μπορούν και οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές τις ε, ε, ενέργειες, όχι σαν εναλλακτική λύση για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά ως συμπλήρωμα. Αλλιώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα δεχόταν ποτέ να υποκατασταθεί από την άμεση δράση των πολιτών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πολίτες να μπαίνουν στο διάλογο σε σχέση με τις πολιτικές και αν η Κομισιόν εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες, ναι, δυστυχώς πολύ συχνά πρέπει να πούμε ότι αυτά τα οποία λένε οι πρωτοβουλίες είναι έξω από τους κανόνες, έξω από τις αρμοδιότητες. Μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες, μπορούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες να κάνουν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Ήδη το έχουμε προσπαθήσει. Έχουμε μιλήσει με αυτούς οι οποίοι κάνουν τις πρωτοβουλίε και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να τροποποιήσουν το περιεχόμενο της ε, πρωτοβουλίας γιατί τότε θα μπει μέσα στους κανόνες. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με αυτούς οι οποίοι αναλαμβάνουν τέτοιε πρωτοβουλίε, αλλά δεν φταίει η Κομισιόν επειδή εφαρμόζει τους κοινώς αποδεκτούς κανόνες θα ήταν πραγματικά σφάλμα να μην εφαρμόσουμε τους κανόνες επειδή μας αρέσει μια πρωτοβουλία. Πρέπει να είμαι λοιπόν στεναρός για το θέμα αυτό. Πρέπει να τονίσω και πάλι ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον κύριο Σέπλουν και τους συνεργάτες τους για να βελτιώσουμε αυτή την ρύθμιση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ακόμα σε αυτό το εργαλείο. Είναι πάρα πολύ εύκολο μετά από τόσο λίγο χρονικό διάστημα να πούμε ότι απέτυχε πρωτοβουλία πολιτών γιατί δεν έχει το χαρακτήρα που θέλετε. Μην μεγαλοποιήσετε το θέμα αυτό, αλλά μην το ακυρώσετε κιόλα τελείω μέχρι ότου έχουμε εξασφαλίσει να λειτουργεί καλύτερα η πρωτοβουλία πολιτών, όπω ζητάει ο κ. Σέφριν και οι άλλοι που υποστήριξαν αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κ. Τίμερμαν. Για να κλείσουμε την συζήτηση, δίνω το λόγο στον κύριο Σέφλιν, τον εισηγητή. Thank you, President. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Όλοι υπήρξαν επικοδομητικοί με μια ή δύο εξαιρέσεις. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τα υποστηρικτικά λόγια του Αντιπρόεδρου Τίμερμανς. Αλλά ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα. Φυσικά δεν μπορώ να συνοψίσω τα όλα όσα υπόθηκαν. Το ζήτημα που ανέφερε ο κύριος Γκέρενς ε, για την αναβάθμιση της δημοκρατικής νομότητας είναι κάτι πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Η σύνδεση των πολιτών αναφέρθηκε πολλές φορές. Το πρόβλημα του follow-up, της παρακολούθησης που αναφέραν πολλοί, ε, ο, ο κύριος Τερικόβιος. Και κάτι άλλο κύριε Τίμπερμανς, κανείς δεν το γνωρίζει αυτό. Εγώ ξέρετε έχω ένα παλιό σκουριασμένο πτυχίο νομικής και ένα από τα πράγματα που έμαθα τότε όσον αφο... είναι ότι όσον αφορά η εφαρμογή των κανόνων πάντα αφήνει κάποιο περιθώριο ερμηνείας. Οπότε θέλω να σας κάνω έκκληση για μεγαλύτερη ευελιξία, για εφαρμογή των κανόνων, αλλά όταν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, ε, μην ξεχνάτε το 1 εκατομμύριο ανθρώπους που υπέγραψαν Τέλο τρία μικρά ζητήματα. Αλλαγή των συνθήκων. Αυτό αναφέρθηκε. Η απόψη μου είναι ναι, η αλλαγή των συνθήκων θα γίνει κάποια ε, μέρα, αλλά όχι βάσει Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Το πρωτεύον δίκαιο δεν εντάσσεται σε όλα αυτά. Δεύτερον, τη στιγμή που γίνεται έκκληση μέσω μια πρωτοβουλίας για να δράσει η Κομισιόν με κάποιο τρόπο, ε, μπορούμε να επαναξετάσουμε την νομοθεσία, τη, διαδικασία αυτή. Από ό,τι κατάλαβα, οι πρωτοβουλίες αυτές δεν μπορούν να επηρεάσουν τρέχουσες διαδικασίες. Ε, οπότε, ε, ξέρετε, οι πολίτες δεν πάβουν να είναι ενδιαφερόμενοι στα πολιτικά ζητήματα της Ευρώπης. Οπότε να ευχαριστήσω τον κύριο Τιμπερμάντ και να πω ότι όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ε, η μπαλά είναι στο γήπεδό σα ε, και είμαι βέβαιο ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να την μετατρέψετε σε μια πολιτική βιώσιμη. Ευχαριστώ κύριε Σέφλιν. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα.